Mes chers collègues, bonjour. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Ζητώ συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση. Κοιτάξτε, είπα καλημέρα σα, διορθώνει η Δερμηνέα. Χάσατε, λέτε ακόμα, λέμε ακόμα καλημέρα και με με διορθώνετε, γιατί καλησπέρα λέμε μετά τι 6 το απόγευμα. Καλημέρα λοιπόν Ισμαήλ, πώς πας, ελπίζω όλοι να είστε καλά. Να εγκριθεί το σχέδιο ημερήσια διάταξης, αν είστε όλοι ικανοποιημένοι και δεν έχετε αντιρρήσεις. Να εγκρίνουμε επίσης και τα πρακτικά της 12ης Απριλίου, εάν δεν υπάρχουν επίσης αντιρρήσεις. Ανακοινώσει τη Προέδρου. Μεγάλη η τύχη σας γιατί δεν υπάρχουν. Ξεκινούμε λοιπόν ευθύ αμέσω. Με ε, τη χρέωση για τη χρήση των ε, δικτύων οδικών δικτύων υποδομής έχουμε την εισηγήτρια, την επιβολή τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομής. Ο κύριος Σαλίνη δεν είναι εδώ ούτε και κάποιοι άλλοι. Χαιρετώ την κυρία Γαϊβόντα Λον Μπονφουά. Δεν ξέρω γιατί υπάρχουν τόσε απουσίε. Τσαγκαρό Δευτέρα μάλλον. Πριν δώσω το λόγο στην εισηγήτρια... Α, υποχωρείτε. Χαίρομαι. Πριν δώσω λοιπόν το λόγο στην εισηγήτρια να καλωσορίσω θερμά την ομάδα των επισκεπτών μας από το Πανεπιστήμιο του Βισμπάντεν. Είναι μια ομάδα φοιτητών νομικής. Σηκώστε το χέρι παρακαλώ για να σας δούμε και να σας χαιρετήσουμε. Ο κύριος Γκάλαχερ τους ε, έχει προσκαλέσει. Είστε πρόσδεκτοι και να είστε πολύ προσεκτικοί, γιατί η δική μας Επιτροπή είναι εξόχως νομοπαρασκευαστική και εσείς που σπουδάζετε νομική ίσως είστε και μελλοντικοί νομοθέτες που θα εργαστείτε σε αυτή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα μάθετε πολλά περνώντας το απόγευμά σας μαζί μας. Ξεκινούμε λοιπόν με το πακέτο τη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα. Να δώσω πρώτα το λόγο στην εισηγήτρια και μετά στους σκιώδεις εισηγητές, τον κύριο Ντάνς, που είναι ο κύριος Ντάνς, δεν είναι εδώ. Η κυρία Κλούν λείπει. Θα ακούσουμε την άποψη της Επιτροπής Ένβη και μετά θα ακούσαμε ε, και τα μέλη της δικής μας Επιτροπής. Πώς πάτε μέλη της Επιτροπής μας Μεταφορών, πώς θα πάτε δύσκολα, γιατί είναι Δευτέρα απόγευμα. Εν πάση περιπτώσει, έχετε το λόγο Κυρία Γαϊβό Νταλόν Μπονφουά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πριν παρουσιάσω τις συμβαστικές τροπολογίες πάνω στις οποίες έχουμε δουλέψει εξαιρετικά πολύ με τους σκιώδεις εισηγητές, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους θερμά για τη συνεργασία σας εντός Επιτροπής μας και μεταξύ των άλλων Επιτροπών και για την ενεργή σας συμμετοχή για τη διατύπωση των συμβαστικών λέξεων. Αναφέρομαι κυρίως στους σκιώδεις εισηγητές, οι οποίοι επέδειξαν καλή θέληση και παρόλο που όλες οι συμβιβαστικές τροπολογίες δεν στηρίζονται από όλες τις πολιτικές ομάδες, λογικό και φυσικό αυτό, καταφέραμε να πετύχουμε την μέγιστη δυνατή συνένεση. Συμβιβαστική τροπολογία για το πρώτο είναι πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε τα έσοδα από τα διόδια ε, να ε, τίθεται κατά μέρος και να μπορούμε να τα αναγνωρίζουμε για τις επιβαρύσεις των διοδίων στις ε, ορεινές περιοχές, για την ε, για την σταθμισμένη διαφοροποίηση των διοδίων ε, σε σχέση με τις περιφέρειες, τις εξόγως απόκεντρες περιοχές ή σε σχέση με το μέγεθος ε, και το πόσο ρηπαίνουν τα βαρέα οχήματα. Όλες αυτές οι διαφοροποιήσεις είναι πολύ σημαντικές. Ε, και χαίρομαι γιατί στις 31 Ιανουαρίου του 2022 τελειώνει και η επιβολή του τέλους κυκλοφορίας από τη στιγμή που θα αντικατασταθεί με τα νέα ε, μέτρα που έχουμε προβλέψει. Και έτσι ε, εφαρμόζουμε και την αρχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο ρηπαίνων πληρώνει και ο χρήστης πληρώνει. Θα έχουμε μια συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών αύριο για να οριστικοποιηθεί αυτή η συζήτηση. Ως προς το τέλος για το εξωτερικό κόστος να υιοθετήσουμε τις ελάχιστες τιμές και αξίες για το ύψος αυτών των τελών σε σχέση με το τι ε, κατάταξη έχουν στο, στην ε, ε, ξυνόμηση γιούρο των οχημάτων. Αυτό προτείνει η Επιτροπή ΕΝΒΗ και σε ό,τι έχει να κάνει με τη συμβαστική τροπολογία για τα τέλη κυκλοφορία για τα ελαφρά οχήματα, χρέον είναι να συνεχιστεί η συζήτηση. Καταλαβαίνω τις ανησυχίες ορισμένων μελών, όμως η 31 Ιανουαρίου του 2025 μας επιτρέπει να έχουμε προοδευτική υιοθέτηση των μέτρων και να έχουν τα κρατημέλη επαρκή χρόνο στη διάθεσή τους για να συμμορφωθούν με το ευρωπαϊκό κανονιστικό νομικό πλαίσιο και για να αποφύγουν αποφύγουμε τις παρεξηγήσεις. Τα τέλη για την κυκλοφοριακή συμφόρηση παραμένουν μη δεσμευτικά το κείμενο δίνει τη δυνατότητα στα κρατημέλη να επιβάλλουν τέτοιου είδου τέλη με εναρμονισμένο τρόπο εφόσον το επιθυμούν. Δεν είναι δεσμευτικό και υποχρεωτικό. Καταλαβαίνω τις επιφυλάξεις ορισμένων βουλευτών και τους καθησυχάζω για τον μη δεσμευτικό χαρακτήρα αυτή του μέτρου. Τώρα για τα δευτερογενή δίκτυα οδικά. Δεν είναι υποχρεωμένα τα κράτη-μέλη να επιβάλλουν διόδια, είναι μια δυνατότητα που μπορούν να επιβάλλουν. Η συμβαστική αυτή τροπολογία έχει να κάνει με το εξή. Αν τελικά τα κράτη-μέλη επιβάλλουν διόδια, τότε να το κάνουν με βάση το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο της σχετικής οδηγίας και να αποφύγουν απλά να μετακυλιστεί η κυκλοφορία σε αυτά τα δευτερογενή οδικά δίκτυα μεταφορών. Συμπερασματικά πιστεύω ότι διατηρούμε το υψηλό επίπεδο φιλοδοξιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενισχύουμε ορισμένα σημεία όπως είναι το τέλος για το εξωτερικό κόστος και βελτιώνουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί λαμβάνουμε υπόψη τον αντίκτυπο που έχει σε επίπεδο δαφικό και κοινωνικό το σύστημα των τηλεδιοδίων. Και να ξέρετε ότι έχουμε και άλλη συνεδρίαση εργασίας αύριο για να προχωρήσουμε έτσι περαιπέρα. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Ζος Μπάρ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα ήδη από την αρχή να αναφέρω ότι είχαμε πολύ καλή συνεργασία με την εισηγήτρια καθώς και με τους άλλους σκιώδεις εισηγητές. Νομίζω ότι η διαδικασία ήταν γενικά ικανοποιητική για όλους. Όπως ε, είπε και η συγγήτρια η Κριστίν, ε, μπορούσαμε να καταλήξουμε σε πολύ καλές ε, συμβιβαστικές τροπολογίες. Το ΕΛΚ δεν μπορεί να συμφωνήσει με τον συμβιβασμό για τα τέλη συμφόρησης, διότι πιστεύουμε ότι έτσι θα έχουμε διπλή επιβάρυνση. Δεύτερο σημείο που δεν μπορεί να στηρίξει το ΕΛΚ είναι η επέκταση των μέτρων ώστε να συμπεριλαμβάνουν και ε, ε, ε, δευτερεύουσες οδούς. Αυτό είναι προαιρετικό. Παρ' όλα αυτά το ΕΛΚ θεωρεί ότι λόγω της επικουρικότητας θα πρέπει να εναπόκειται στα κράτη-μέλη να αποφασίσουν ποιες δευτερεύουσες οδοί θα καλύπτονται διότι γνωρίζουν καλύτερα. Πιστεύουμε ότι δεν ε, είναι χρήσιμο να έχουμε ενιαίο κανόνα για όλους. Όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων, πιστεύουμε ότι μπορέσαμε να καταλήξουμε σε καλή συμβιβαστική πρόταση. Στο μέλλον έτσι θα έχουμε πολλά δεδομένα στη διάθεσή μας ε, χωρίς να δημιουργήσουμε ένα γραφειοκρατικό τέρας, κάτι που θέλουμε να αποφύγουμε. Επίσης ε, χαίρομαι που πετύχαμε ευρεία πλειοψηφία υπέρ ε, του συμβιβασμού για τα μικρά, τα ελαφρά φορτηγά. Το θέμα των θέσεων στάθμευσης ε, επίσης καλύπτεται κάτι το οποίο βρίσκω επίσης πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι έχουμε δύο ακόμα θέματα που ανέφερε η συγγήτρια. Την ε, βαθμιαία κατάργηση για τα επιβατηγά. Θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό και ένα ακόμα θέμα που θα πρέπει να συζητήσουμε είναι ο διαχωρισμός ε, των λεωφορείων και των φορτηγών. Ε, προσβλέπω στην ε, συζήτηση των σκιωδών εισηγητών αύριο και ελπίζω να μπορέσουμε να υιοθετήσουμε μια καλή έκθεση τελικά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπάρα. Κύριε Ρικέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την εισηγήτρια για την ποιότητα της δουλειάς της, των προκατακτικών εργασιών καθώς και των συζητήσεων. Η θέση της ομάδα μας γενικά δεν ήταν πολύ διαφορετική. Οι συζητήσεις λοιπόν δεν ήταν δύσκολες. Συμφωνούσαμε με την ιδέα ότι έπρεπε να επερβούμε την πρόταση, το πλαίσιο της πρότασης της Κομισιόν και να επιτύχουμε κάποιες ε, θέσεις ε, ε, ε, ε, Ξέρουμε βέβαια το earmarking ε, ξέρουμε ότι θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα σε πιθανό τρίλογο, αλλά το υποστηρίζουμε. Επίσης και για τα επαγγελματικά οχήματα την επέκταση συμφωνούμε. Για το πρόβλημα των δευτερευουσών οδών Συμφωνούμε με την εισηγήτρια ότι αυτές οι δευτερεύουσες οδοί πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε περίπτωση που προβλεφθεί ε, σε αυτό το κανονισμό. Γιατί, διότι αν δεν συμπεριληφθούν, να τις παρακάψουμε ε, με αιτιολογία την επικουρικότητα, αυτό θα δημιουργήσει κινδύνους για την εσωτερική αγορά. Αν βρούμε δηλαδή παρακαμπτήρες λύσεις ε, που δημιουργούν πρόβλημα ε, γεωγραφικό και διοικητικό ουσιαστικά. Δεν πρέπει λοιπόν ε, να μας εμποδίσει αυτό από τη γενικότερη εφαρμογή της, ε, του κανονισμού από ότι υποστηρίζουμε τη θέση της συζυγήτριας. Κάτι άλλο σημαντικό για την ομάδα μου είναι η δυνατότητα οι περιφερειακέ αρχέ με την επιφύλαξη τη Συμφωνία των Κρατών Μελών να μπορούν να ρυθμίσουν κάποια πράγματα. Αυτό σχετίζεται και με το ζήτημα των δευτερεύουσων οδών. Πολύ συχνά, πέραν των μεγάλων δικτύων, ε, οι περιφερειακές αρχές είναι οι καλύτερες. Είναι αυτές που μπορούν καλύτερα στο πλαίσιο αυτής της οδηγίας ε, να αποφασίσουν ενδεχομένω ε, εφαρμογή τυχών τελών για τα ασφαλείς χώρους στάθμευσης όλοι αντιλαμβάνονται πόσο σημαντική είναι φυσικά κυρίως για άλλους κανονισμούς αλλά δεν μπορούμε να τους συσχετίζουμε με τις έννοιες των αυτοκινητοδρόμων συστηματικά. Δεν πρέπει να έχουν αυτόν τον υποχρεωτικό χαρακτήρα ε, όσον αφορά την εφαρμογή αυτής της οδηγίας γιατί ε, έτσι τα πράγματα θα ήταν μη διαχειρίσιμα όπως έχουν τα πράγματα σήμερα. Δυστυχώ στου μεγάλου έξονε ε, δεν έχουμε ακόμα τέτοιου χώρου, δεν έχουν επιληθεί ακόμα όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με την εκμετάλλευση, όχι μόνο με την επένδυση, αλλά και με την εκμετάλλευση των χώρων αυτών στάθμευση. Η αρχή λοιπόν του να πληρώνει ε, της ε, κατά απόσταση. Το earmarking είναι οι τρεις βασικοί πυλώνες του, κανόνα αυτού, του κανονισμού αυτού. Ε, τους υποστηρίζουμε. Δεδομένου των αντιδράσεων που έχουμε αντιληφθεί εκτός του Κοινοβουλίου, όπως φαντάζεστε, οι συζητήσεις με το Συμβούλιο θα είναι δύσκολες. Η ευρεία συνένεση λοιπόν που πέτυχε η συγγήτρια θα αποδειχθεί εξαιρετικά ωφέλιμη για τις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν, ε, οι οποίες θα είναι δύσκολες. Από την ομάδα μας θα υπάρχει ευρία υποστήριξη πάντως ε, και έχουν βρεθεί και σχετικά με αυτό πολλές ε, συμφωνίες, πολλοί συμβιβασμοί. Ευχαριστούμε κύριε Ερικέ, κύριε Ντελάντερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ο συνάδελφος ε, Μίχαελ Κράμερ που είναι αρμόδιος για το θέμα αυτό δεν μπόρεσε να είναι παρόν. Γι' αυτό θα πω λίγα λόγια εκ μέρους του. Βλέπουμε πολλές ε, θετικές πτυχές ε, στην πρόταση αυτή. Μεταξύ άλλων το ότι θέλουμε να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογή ώστε να συμπεριληφθούν και οι δευτερεύουσε οδοί. Επίσης τα τέλη να βασίζονται στην απόσταση και να έχουμε και ελάχιστε αξίε. Πιστεύουμε ότι αυτά είναι πολύ θετικά. Ε, διότι πιστεύουμε ότι θα πρέπει να έχουμε εξωτερικοποίηση του κόστους με συμπερίληψη του κόστους ε, για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Ε, κάποια θέματα που μας λείπουν είναι να συμπεριλαμβάνονται ιοταχή και μοτοσικλέτες για να καλύψουμε το σύνολο του τομέα μεταφορών, αλλά επίσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να συμβάλλει στην εφαρμογή αυτών των ε, μέτρων. Η πρόταση αυτή λοιπόν έχει και καλά ε, σημεία και λιγότερο καλά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κυρία Κιλόνεν, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία ε, εσάς κυρία εισηγήτρια, αλλά και τους κοιόδες εισηγητές να ευχαριστήσω. Πράγματι λοιπόν, είναι απολύτως απαραίτητο να σημειώσουμε πρόοδο σε ό,τι έχει να κάνει το τομέα των μεταφορών και να βελτιώσουμε την κατάσταση της υγείας όλων βελτιώνοντας τον τομέα των μεταφορών. Η συνάδελφος έκανε μια πολύ επικοδομητική δουλειά και έχει υποβάλει μια σειρά από προτάσεις. Πρέπει να πω ότι είμαι ικανοποιημένη με τις ε, συμβιβαστικές τροπολογίες. Θα θέλαμε ίσως μια κάποια κάπως διαφορετική διατύπωση σε θέματα ασφάλειας, μεταφορών, υποχρεώσεων. Είμαστε έτοιμοι και να συζητήσουμε για την κατάσταση που έχει να κάνει με τα λεωφορεία και τα φορτηγά. Να οριστικοποιήσουμε κάποιες λεπτομέρειες. Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά θεωρώ ότι μπορούμε να τα στη συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών. Ποιος είναι ο στόχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχει να κάνει με το, την Ευρωβινιέτα, με το Ευρωπαϊκό Τέλος Κυκλοφορίας, με το περιβάλλον, Ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Ένας τριμερής διάλογος θα μας οδηγήσει κάπου όπου θα υστερούμε σε σχέση με αυτό που ζητά από μας το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Ας ελπίσουμε ότι η απόσταση δεν θα είναι πολύ μεγάλη. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ για τη συνεργασία και για το επικοδομητικό πνεύμα. Θα τα δούμε όλα αυτά αύριο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Αγίου το παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια. Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Την παρακολούθησα και είδα και τα συμπεράσματα. Είμαι βέβαιη ότι θα καταλήξουμε σε ένα κείμενο το οποίο θα μας βρει στο μέγιστο βαθμό όλους σύμφωνους. Όσον αφορά εμένα προσωπικά, επιβεβαιώνω τις θέσεις που έχω ήδη εκφράσει πλήρη υποστήριξη στην αρχή του «Ο χρήστης πληρώνει και ο ρήπανον πληρώνει». Οι προβληματισμοί επιφυλάξεις που παραμένουν αφορούν το δευτερεύον δίκτυο. Παρότι στη διατύπωση που προτείνεται στη συμβιβαστική πρόταση το όραμα που υπάρχει μας βρίσκει περισσότερο σύμφωνο σε σχέση με τις αρχικές θέσεις, διότι αντιλαμβάνουμε ότι σε ορισμένε χώρες το επίπεδο των δευτερευουσών αποδομών ε, είναι συγκρίσιμο με αυτό των πρωτευουσών, οπότε αυτή η συζήτηση ε, που επιθυμούσε η εισηγήτρια αιτιολογείται πλήρως. Αλλά σε άλλα κράτη-μέλη οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου, υπερβολικά μεγάλες ακόμα. Οπότε το να αφήσουμε την ελευθερία, την πρωτοβουλία στα κράτη-μέλη να αποφασίσουν να εφαρμόσουν ή όχι τέλη στο δευτερεύον δίκτυο είναι και αυτό μια πρόταση. Ε, εκεί όμως θα είναι δυσανάλογα τα αποτελέσματα. Όσον αφορά τα κίνητρα και τις εξαιρέσει για τα οχήματα μηδενικών εκπομπών, είμαστε απόλυτα υπέρ, διότι ούτως ή άλλως κάτι πρέπει να κάνουμε για να υπάρξει ε, σωστά αυτή η μετάβαση στη χρήση ε, λίγο, οχημάτων που ρηπαίνουν λιγότερο. Αλλά όπως οποιοδήποτε κίνητρο και σχετική στήριξη δεν μπορεί να διαρκέσει για πάντα. Θα πρέπει να εφαρμοστεί δια... με κάποια διαβάθμιση ευθύνουσα. Οπότε θα πρέπει να δούμε ποια οχήματα και όσο θα αυξάνει το αριθμός τους ε, να αλλάζει το τέλος. Η πόροι επενδύονται για να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία. Δεν μπορούμε να προσφέρουμε τέτοια στήριξη επάπειρων. Στο σύνολο συμφωνούμε με την πρόταση. Η πρωτοβουλία Ε, να υπάρχουν παρόμοια τέλη με του σιδηροδρόμου στι οδικέ μεταφορέ. Συμφωνούμε. Αλλά κάποιε κατηγορίε πρέπει να προστατευτούν. Οι άνθρωποι που ταξιδεύουν καθημερινά για να πάνε στη δουλειά του, οι άνθρωποι χαμηλών εισοδημάτων. Πρέπει δηλαδή να δώσουμε ε, κάποια ευκολίε για τους πολίτες. Οι πολίτες αυτοί θα πρέπει να μπορούν να επαληθεύσουν ε, ότι πράγματι υπάρχει κάποια επένδυση ορατή σε υποδομές και σε συνθήκες ασφαλείας. Αλλιώς απλά τους αυξάνουμε το κόστος. Οπότε ας προσπαθήσουμε να μην τιμωρούμε κανέναν, να είναι ορατές αυτές οι επενδύσεις, να φαίνονται στις υποδομές. Κατά τα άλλα, να επαναλάβω, στο σύνολο υποστηρίζουμε την πρόταση και αναμένουμε να δούμε σύντομα το τελικό κείμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Γιώτο, κυρία Αρνότου, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία εισηγήτρια για τη δουλειά σας. Ας μην χανόμαστε σε περί τα πράγματα. Όποιοι συμβαστικές και να πετύχατε κύριε εισηγήτρια, η αλήθεια είναι ότι τα κράτη που στις πιο πλουσιές υπήρου του πλανήτη δεν έχουν τα μέσα μετά από 20 χρόνια λιτότητας να συντηρήσουν τις οδούς τους ε, ισχυριζόμενοι τώρα ότι προφυλάσσουμε το περιβάλλον λέμε να αντλήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα από του οδηγού γιοταχή, ενώ στην αρχή η έκθεση αφορούσε μόνο τα βαρέα οχήματα. Και έτσι η έκθεση αυτή έγινε ένα μέσο ώστε να αρμέξουμε όσο το, δυνατότερο, περισσότερο δυνατό του οδηγού στην γιοταχή. Ε, να έπρεπε να έχουμε αυτή τη φορολόγηση των βαρέων οχημάτων που θα έπρεπε να πληρώνουν για τις οδούς που χρησιμοποιούν όλοι συμφωνούμε σε αυτό, κανείς δεν το αμφισβητεί ακόμη και μεγαλύτερες ε, μεταφορικές ε, που απλά συζητούν τις προϋποθέσεις τώρα εγώ ως αιρετή του γαλλικού λαού δεν θα συμμετέχω σε αυτό το πονηρό παιχνίδι θα καταψηφίσω λοιπόν όλες τις τροπολογίες και τις συμβιβαστικές συμπεριλαμβανομένων κυρίως αυτές τις εισηγήτριες που κατ' εμέ αυξάνουν απλά τα τέλη για τους οδηγούς. Να υπενθυμίσω τέλο για όλου ισχυρίζονται ότι υποστηρίζουν την ελευθερία, ότι μια τη πρώτη ελευθερίε είναι η ελευθερία ε, κυκλοφορία. Δεν μπορούμε λοιπόν να την περιορίζουμε ε, ανάλογα με τα οικονομικά μέσα των πολιτών. Ευχαριστώ. Ωραία. Συνεχίζουμε, κυρία Κόρντ. Ο κύριος Κοχ, αγαπητή Κριστίνε, ε, χαίρομαι πολύ με τις ε, γενικά εξαιρετικές ε, συμβιβαστικές τροπολογίες. Παρ' όλα αυτά κάποιες παρατηρήσεις. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με καμία συμβιβαστική πρόταση που να επιτρέπει έστω και προαιρετικά τέλη συμφόρησης. Πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε διπλή επιβάρυνση. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να καταργηθούν τα τέλη συμφόρηση και να μην ε, εισαχθούν νέα. Δεύτερον, τα κράτη-μέλη θα έχουν την ε, δυνατότητα αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος ε, που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 παράγραφος 7 να μπορούν να τα να τα συμπεριλάβουν. Και μιλάμε για ιστορικά ε, πολύτιμα οχήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κόχ. Κύριε Σμιτ, παρακαλώ έχετε το λόγο. Ε, σας ευχαριστώ πολύ και εγώ πιστεύω ότι έχει γίνει εξαιρετική δουλειά από πλευράς της εισηγήτριας και από πλευράς των σκιωδών εισηγητών που ε, δεν ήταν δύσκολο να συμβιβάσουμε τις προτάσεις μας. Ε, στον συνάδελφο Νταλούντε να πω ότι δεν ε, θέλουμε εδώ μια θετική πράσινη μεταρρύθμιση, θέλουμε μια λογική λύση για τους οδηγούς της Ευρώπης. Ε, διαφωνώ με τα τέλη συμφόρησης. Έτσι γίνεται πολύ πιο ακριβή η οδήγηση σε αυτοκίνητο και επίσης, όπως είπε ο συνάδελφος, αντίκειται στην αρχή της επικουρικότητας που θεωρώ ότι είναι μία από τις σημαντικότερες. Επίσης, ε, η προοδευτική δομή ε, των ε, τελών δεν έχει κανένα νόημα, διότι το κόστος δημιουργίας των οδών μπορεί να γίνει μέσω των τελών των ορυκτών καυσίμων. Επίσης, ε, δεν χρειάζεται να έχουμε ευρωπαϊκό σύστημα διοδίων που να βασίζεται στην απόσταση. Η οδηγία ε, για την ε, Ευρωβινιέτα στόχο είχε να αντιμετωπίσει τις ανισότητες στον αντιγωνισμό. και ε, σε διάφορες διαδρομές δεν υπάρχει και ανταγωνισμός ουσιαστικός όταν εγώ παίρνω το αυτοκίνητό μου. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναπόκειται στα κράτη-μέλη να ε, αποφασίσουν πώς θα διαμορφώσουν τα τέλη των διοδίων. Και βέβαια ε, διάκριση με βάση την εθνικότητα, την υπηκότητα των οδηγών δεν επιτρέπεται καθόλου να γίνει. Επίσης, ε, τα τέλη συμφόρησης... Ε, για τα τέλη συμφόρηση θα ήθελα να πω το εξή. Κανεί δεν θέλει να κολλήσει στην κίνηση και πολλοί, δεν, ε, πολλοί επαγγελματίε δεν μπορούν να επιλέξουν την ώρα που θα χρησιμοποιήσουν τους δρόμους. Είναι απλά μια ακριβή παρενόχληση και δεν νομίζω ότι επιτρέπεται η Ευρώπη να κάνει τέτοια πράγματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δελίλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω δύο σύντομες παρατηρήσεις να κάνω. Σημεία στα οποία μας εφίστησε την προσοχή ως και εισηγητής κύριος Τζόρτζ Μπαχ. Μιλούμε για την επιβατική μεταφορά σε πούλμαν και ελοφορία συμβάλλουν τα μάλλα στη μείωση της κυκλοφορίας και στη μείωση των εκπομπών. Δεν είναι όμως τόσο διαδεδομένος αυτός ο τρόπος μεταφοράς σε όλα τα κράτη-μέλη. Η παρουσία αυτού του δικτύου συσχετίζεται με την παρουσία συνδροδρομικού δικτύου και προσβασιμότητα σε αυτά. Θεωρώ λοιπόν ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να διατηρήσουν αρκετή ευελιξία για να προσωποποιήσουν την προσέγγισή τους στις δικές τους ανάγκες όταν πρόκειται για την επιβολή τελών σε πούλμαν και ε, λεωφορεία ε, μεταφοράς επιβατών. Τώρα για τα επιβατικά οχήματα θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί και να αφήσουμε τα κράτη-μέλη να διαλέξουν εκείνα το πιο αποτελεσματικό ε, τρόπο επιβολής χρέωσης. Κανείς δεν αμφισβητεί την αρχή ο ρηπαίνων πληρώνει και ο χρήστης πληρώνει. Αλλά δεν είναι τρόπος να προχωρήσουμε με υποχρεωτική εφαρμογή. Οι πολίτες απλά θα αλλάξουν ε, τους δρόμους που χρησιμοποιούν, θα χρησιμοποιούν πιο επαρχιακούς, πιο δευτερεύουσε οδούς και θα δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερη συμφόρηση ε, και ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή επικουρικότητα και ευελιξία. Αυτό είναι αυτό που πρέπει να διατηρήσουμε στον τρόπο επιβολής τελών των επιβατικών οχημάτων. Αυτό είναι στοιχείο κλειδί για την επιτυχία αυτού του φακέλου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριος Λιμπεράτσικη παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ την Κατρίν, την εισηγήτρια, ήταν πολύ δύσκολο να καταλήξει στη λύση που έχουμε μπροστά μας. Επομένως, θεωρώ ότι επειδή έχουμε ένα τέλος εποχής αυτή τη στιγμή, ε, Χρειαζόμαστε όλο και περισσότερους δρόμους. Ο χώρος όμως είναι πεπερασμένος και θέλουμε οι δρόμοι να χρησιμοποιούνται όσο δυνατό περισσότερο. Το πρόβλημα είναι η διαθεσιμότητα και οι τιμές αναλόγως με την ιδεολογική σκοπιά από την οποία βρίσκεται κανείς. Ε, αυτό είναι το όνομα του παιχνιδιού και τα σημεία των καιρών, τούτων λεχθέντων. Εστρέφουμε προς την εισηγήτρια και θέτω υπόψη της το εξής. Εάν επιβάλλουμε διόδια στις δευτερεύουσες οδούς, τότε δεν θα έπρεπε να έχουμε μια σειρά συστάσεων έτσι ώστε τα χρήματα να ε, τεθούν κατά μέρος για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας αυτών ακριβώς των δευτερεύουσων οδών και κυρίως τα σταυροδρόμια εκεί όπου συναντώνται με ε, τους σιδηροδρόμους. Οι σιδηρόδρομοι δεν επενδύουν γιατί λένε ότι πρέπει αυτοί που ασχολούνται με τις οδικές μεταφορές να επενδύσουν στο σταυροδρόμι. Και ο φορέας εκμετάλλευσης, η εταιρεία που έφτιαξε το δρόμο, λέει δεν είναι δικιά μας δουλειά και ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Όλο και περισσότερα είναι τα ατυχήματα μεταξύ οχημάτων και τρένων. Πρέπει λοιπόν να αναπτύξουμε τους σιδηροδρόμους και κάποια από τα χρήματα που εισπράττουμε να τα θέσουμε κατά μέρος και να τα αφιερώσουμε στην ενίσχυση των επενδύσεων για να προστατεύσουμε ε, τα σημεία διάσχησης από τα αυτοκίνητα των σιδηροδρομικών γραμμών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ομιλήτρια παρακαλώ. Η κυρία Κράσβαντερ Χάιν, ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε. Τα εξωτερικά κόστη θα πρέπει να συμπεριληφθούν, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη μας ε, και ε, τις ε, ουσίες στην ατμόσφαιρα. Στην Αυστρία έχουμε ένα σύστημα βινιέτας. Δεν θα είναι πρόβλημα λοιπόν για μας το να υπάρχει το να μην υπάρχει ευρωπαϊκό σύστημα, διότι το να εισαχθεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα διαφορετικό από αυτό που έχουμε εμεί στην Αυστρία θα σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε μεγάλε αλλαγέ στην Αυστρία. Δεν ε, θέλουμε να ε, εκχωρήσουμε το πρότυπο αυτό που χρησιμοποιούμε ήδη. Ε, δεν καταλαβαίνω ακριβώς πώς θα διαμορφωθούν τα μέτρα αυτά. Ε, αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, ε, πρέπει να ε, ε, επανεπεξεργαζόμαστε την πρόταση για τι Χρειαζόμαστε όμω και ένα ενιαίο σύστημα διοδίων στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Στρέφομαι προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Εντιλιζό. Έχετε το λόγο. Θα ήθελα να επιμείνω σε κάτι που νομίζω ότι είναι σημαντικό όταν συζητάμε την Ευρωβινιέτα όταν νομοθετούμε στην Επιτροπή Μεταφορών γιατί έχουμε κάποιους στόχους. Ένας από τους μείζονες στόχους είναι μια πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και επειδή ουσιαστικά χορεύουμε μέσα σε ένα ηφαίστειο, όπως λέει η Πρόεδρος, ε, κλιματική, τις κλιματικές δυσκολίες, ε, δεν πρέπει να παραβλέπουμε και την δημόσια υγεία. Είναι τεράστια τα νούμερα στην Ευρώπη. 500.000 πρόωροι θάνατοι, το υπενθυμίζω. Οπότε, αν μπορέσουμε να ψηφίσουμε κάτι το οποίο θα βοηθήσει στην καλή υγεία των συμπολιτών μας θα ήταν καλό. Παρακαλώ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν μου επιτρέπετε δύο παρατηρήσεις προκαταρκτικές επί του συνόλου των εκθέσεων. Να σημειώσω πρώτα απ' όλα ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν γίνει πολλές συζητήσεις και συνεδριάσεις με την εισηγήτρια του Σκιώδους, τη γραμματεία της Επιτροπής σας, πολύ επικοδομητικές και θετικές συζητήσεις. Και σήμερα θα ήθελα να το επισημάνω αυτό και να σας ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές για την πολύ θετική σας στάση. Το δεύτερο μήνυμα που ήθελα να δώσω γενικά αφορά το χρονοδιάγραμμα, το timing. Όπως ξέρετε, οι συζητήσεις στο Συμβούλιο δεν είναι εύκολες. Στις 7 Ιουνίου θα έχουμε ένα Συμβούλιο Υπουργών και εκεί ελπίζουμε να καταλήξουμε σε μια γενική προσέγγιση. Σε αυτό το δυσχερές πλαίσιο πρέπει να πω. Εδώ έχει το Κοινοβούλιο πιστεύω να παίξει σημαντικό ρόλο σίγουρα επί της ουσίας αλλά εξίσου και σε θέματα χρονοδιαγράμματος. Θέλουμε λοιπόν να ενθαρρύνουμε την Επιτροπή Τραν να υιοθετήσει, να κλείσει τις εκθέσεις στο δικό της επίπεδο το συντομότερο δυνατόν, εφόσον αυτό είναι δυνατόν. 24 Μαΐου όπως είχε προβλεφθεί ή σε κάθε περίπτωση πριν από, την, από το Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της 7ης Ιουνίου ώστε να δώσουμε ένα μήνυμα ότι κινούμαστε προς αυτό στο να κλείσουν τα μεγάλα θέματα πριν από το τέλος αυτής της εντολής. Αυτές είναι οι γενικές μου παρατηρήσεις. Όσον αφορά αυτή την έκθεση που αφορά την τρίτη αναθεώρηση της οδηγίας για την Ευρωβινιέτα, είναι ένα όνομα μόνο η Ευρωβινιέτα. Απέχουμε πολύ από την οδηγία που υιοθετήθηκε πριν από πάνω από 20 χρόνια. Ήταν μια φιλόδοξη πρόταση της Επιτροπής τότε για τα ε, οχήματα που καλύπτονταν για τα εξωτερικά κόστη και πρέπει να πούμε ότι η κυρία Ρεβόνταλόν είναι ακόμη πιο φιλόδοξη. Βρίσκεται, πιστεύω, στην ίδια γραμμή με τις λευκές βίβλους της Κομισιόν και όσον αφορά την υλοποίηση των αρχών του ορυπαίνων και ο χρήστη πληρώνει. Όπω ξέρετε, σε επίπεδο Συμβουλίου, δυστυχώ οι εργασίε δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Σήμερα το πρωί συναντηθήκαμε με την Αυστριακή Προεδρία που έχει πρόθεση να ξεκινήσει τις εργασίες ε, το πακέτο για την κινητικότητα. Σίγουρα αποτελεί πρωτοβουλία για την Αυστριακή Προεδρία για όλα τα θέματα για τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσει, αλλά και για το θέμα του ευρωπαϊκού τέλους κυκλοφορία τη Ευρωβινιέτας. Σίγουρα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο το Κοινοβούλιο πρέπει οπωσδήποτε να υιοθετήσει μια ισχυρή και σαφή θέση όσον αφορά τι αρχές που θέλετε να συμπεριληφθούν σε αυτή την αναθεώρηση τη οδηγία για την Ευρωβινιέτα. Δεν θα μπω στι λεπτομέρειες όλων των ε, σχεδίων τροπολογιών ε, που έχουμε επισημάνει ήδη στι δύο προηγούμενε συζητήσει. Η Κομισιόν θέλει να εκφράσει την υποστήριξή τη γενικά ε, στι εργασίε που έχουν γίνει Επίσης θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι εξαιρετικά υψηλής τεχνικής ποιότητας ε, οι τροπολογίες που έχουν προταθεί από την κυρία Ρεβονταλόν. Μία παρατήρηση, ένα μικρό προβληματάκι που έχουμε επισημάνει σε προηγούμενες ε, παρεμβάσεις μας. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο όταν ε, θέλουμε να φτιάξουμε ένα νέο διόδιο ένα νέο τέλος ε, ή ένα επιπλέον αυτών που ήδη υπάρχουν, θα πρέπει να υπάρχει μια ειδοποίηση προς την Κομισιόν, γιατί ένα τέτοιο μάρκα μπορεί να αποτελεί πολύ μεγάλη αύξηση του βασικού τέλους διοδίων. Γιατί τέτοια ειδοποίηση, όχι γραφειοκρατικά, απλά διότι είναι απαραίτητο να είμαστε βέβαιοι ε, ότι είναι δίκαια το τέλος διοδίων για τους χρήστες. Αυτό θέλουμε να ελέγχουμε. Οπότε θέλουμε να επιθυμήσουμε αυτό στην κυρία εισηγήτρια να μην χορηγήσει επιπλέον εξαιρέσει ε, σε σχέση με την σημερινή οδηγία όσον αφορά τις υποχρεώσεις ε, ε, κοινοποίησης των σχεδίων τελών διοδίων στην Κομισιόν. Μια χώρα που γνωρίζετε πολύ καλά και που προβλέπει ένα markup μετά από πολλές συζητήσεις η χώρα αυτή θα κοινοποιήσει την Κομισιόν, στην Κομισιόν τόσο το συμπληρωματικό τέλος όσο και το βασικό τέλος διοδίων κάτι που θα αποτελέσει εγγύηση για τους χρηστές ότι το τέλος αυτό διοδίων αντιστοιχεί στα, ε, στα όσα προ, ε, η οδηγία. Αυτά για να κλείσουμε πολύ θετικά να σας ενθαρρύνω να προχωρήσετε όσο το δυνατόν συντομότερα για αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε κύριε Λεζόα. Ξαναδίνω το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Κριστίν Ρεβονταλόν. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα ήθελα να πω ότι ψηφίσαμε με συντριπτική πλειοψηφία την αναθεώρηση της Λευκής Βίβλου για τις μεταφορές και αυτή τη διπλή αρχή του ο Ριπένο πληρώνει και ο χρήστης πληρώνει. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που απέχουν οι επόμενες εκλογές σε λιγότερο από ένα χρόνο, ε, ε, σε ένα, χρόνο. Οπότε εδώ πρέπει να δείξουμε ότι ε, τηρούμε τις δεσμεύσεις που είχαμε λάβει και αυτή η έκθεση όπως και άλλες εκθέσεις της Επιτροπής μας είναι το αποτέλεσμα των όσων είχαμε ορίσει εμείς ως αρχές. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ τους συζητητές ε, για τα σχόλιά τους. Όπως βλέπουμε, τα όσα ακούσαμε αφορούν τις συμβιβαστικέ τροπολογίες, οι οποίες ακόμα βρισκόνται υπό συζήτηση. Αυτό που ακούσαμε για τα τέλη συμφόρησης ε, Αντιλαμβάνομαι ότι δημιουργούν κάποιες δυσκολίες για μια-δυο ομάδες. Παρ' όλα αυτά η πλειοψηφία των ομάδων υποστηρίζει αυτές τις προτάσεις και ήθελα να υπογραμμίσω αυτό υπάρχει ήδη σε κάποιες χώρες όπου υπάρχει διαφοροποιημένη χρέωση ανάλογα με την κυκλοφορία της κάθε περιοχής. Είναι κάτι απολύτως κατανοητό και αποδεκτό εφόσον δοθούν οι σωστές εξηγήσεις. Η πρόταση λοιπόν αυτή που προήλθε από την Κομισιόν έχει ήδη αποδειχθεί ε, ότι λειτουργεί σωστά και βοηθά στη μείωση της κυκλοφορικής συμφόρησης και συνεπώς της ρήπανσης. Υπάρχει πάντα αυτή η ιδέα από πίσω. Σε αυτή την ιδέα βασίζεται. Δεν είναι κάτι άλλο πρόσαλο που μας κατέβηκε από το πουθενά. Ε, καταλαβαίνω φυσικά και όπως κατάλαβα ε, το εφαρμόζει και κάποια χώρα σε κάποιους αυτοκινητοδρόμους η χώρα που αναφέρατε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως είπα, δεν θέλουμε να ε, για τις δευτερεύσεις οδούς. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε τέλος διόδιων σε όλες τις δευτερεύσεις οδούς, αλλά όσα κράτη-μέλη το επιθυμούν, τηρώντα την αρχή της επικουρικότητας, μπορούν, δεδομένου ότι ορισμένε δευτερεύσεις οδοί στην πραγματικότητα χρησιμοποιούνται ως παράκαμψη ε, ώστε να αποφεύγουν τα τέλη διόδιων. Και όπω είπε πολύ σωστά ο κ. Λιμπεράτ, και αυτέ οι δευτερεύουσε οδοί που χρησιμοποιούνται ω παρακαμπτήριε για να γλιτώσουν ε, από τα διόδια τίθεται θέμα ασφαλεία. Οπότε για να απαντήσουμε στο τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να υπάρχει ασφάλεια σε αυτέ τι δευτερεύουσε οδού, στι οποίε θα μπορούσαμε να επιβάλλουμε τέλη διοδίων, με ε, θα μπορούσαμε να δώσουμε ως κίνητρο αυτή την ε, δρομολόγηση, όπως είπαμε, των εσόδων. Ε, αυτό μπορεί να οδηγήσει στην αποδοχή του τέλους αυτού. Ε, όπως και οι χρήστες άλλων τρόπων μεταφοράς πληρώνουν για τη χρήση και για τις αποστάσεις που διανύουν. Ακόμα σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι παντού, υπάρχει μια εξαίρεση για τα γεωταχή, για τα ελαφρά οχήματα αυτό υπάρχει σε πολλές χώρες. Οπότε υπάρχει μια ανισότητα σήμερα και η πρόταση που γίνεται εδώ είναι μια πρόταση εναρμόνισης. Δηλαδή όλοι οι τρόποι μεταφοράς συμπεριλαμβάνουμε και του αυτοκινήτου γιατί και εμείς εδώ εκπροσωπούμε τους πολίτες, όχι μόνο τους οδηγούς, γιοταχή, ε, παρότι φανταζομαι ότι όλοι μας οδηγάμε γιοταχή, είναι... Ε, λαμβάνουμε υπόψη ουσιαστικά αυτό, το, το πώς χρησιμοποιείται το αυτοκίνητο σε όλες τις χώρες, ναι, ρηπαίνει και θέλουμε να δούμε ε, τα έσοδα που προκύπτουν από αυτά τα διόδια, πώς θα επανέλθουν στις μεταφορές, ώστε να λαμβάνουμε υπόψη και όλα τα οχήματα, αλλά και τα έσοδα αυτά να επανεπενδύονται στις μεταφορές. Τώρα, όσον αφορά τη διαφοροποίηση μεταξύ των πούλμαν, των λεωφορείων, των φορτηγών, έχουμε κάνει μια διαφοροποίηση στο επίπεδο του τέλους όσον αφορά τα πολυμά και τα λεωφορεία ώστε να λαμβάνουμε υπόψη ότι πρόκειται για μια δημόσια υπηρεσία. Δεν, μπορεί να, δεν μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε ε, όπως τα φορτηγά. Το λάβαμε λοιπόν υπόψη. Άκουσα και τη λέξη tax φόρη. Δεν είναι φόρη, είναι εισφορές στα γαλλικά και το έχω επαναλάβει και άλλες φορές. Το λέω, ότι υπογραμμίζω τέσσερις φορές θα υπάρχει αυτή η αναδρομολόγηση, η επανεπένδυση των εσόδων στις μεταφορές. Είναι κάτι καινούριο. Ε, το έχω υπογραμμίσει πολλές φορές. Αλλά όπως είπε και η κυρία Δέλη και ο κύριος ε, Ρικέ, ε, θέλουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιδείξει δύναμη σε αυτό το θέμα, ώστε πραγματικά να σημειώσουμε κάποια πρόοδο σε αυτό το σύστημα και πραγματικά να γίνει κατανοητό και αποδεκτό το ότι θεσπίζεται εδώ. Αυτό είναι σημαντικό και στον τριμερή διάλογο θα πρέπει να δείξουμε ότι υπάρχει η συντριπτική πλειοψηφία, η ισχυρή πλειοψηφία. Αυτό σα ευχαριστώ. Ραντεβού αύριο για τον τελευταίο μα τριμερή διάλογο επί του θέματος αυτού και δράτω με τις ευκαιρίες για να ευχαριστήσω και τον βοηθό μου Σαμιλ Μπελέ που εργάστηκε σκληρά με όλου μα για την έκθεση αυτή. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι πολύ σαφή όσα μας είπατε. Σας υπενθυμίζω ότι η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στις 24 Μαΐου από τις 9 το πρωί. Συνεχίζουμε λοιπόν με την έκθεση της κυρίας Κλούν, η οποία δεν είναι εδώ. Ο κύριος Βιμ Βαντερκάμ θα την αντικαταστήσει και θα μας μιλήσει για αυτό το θέμα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συνάδελφος Διέντρε Κλούν δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας σήμερα το απόγευμα και θα ήθελα να διαβάσω το κείμενό της. Το δικό της κείμενο και η δική μου ερμηνεία. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για όλες τις τροπολογίες. Εδώ είναι το εύκολο κομμάτι. Λόγω του σχετικά μικρού αριθμού τροπολογιών που δεν ξεπερνά τη 40, δεν θεωρήσαμε ότι είναι απαραίτητο να συντάξουμε συμβαστικές τροπολογίες. Επομένως, πάμε κατευθείαν στη ψηφοφορία και στον κατάλογο ψηφοφοριών. Ως προς το περιεχόμενο, θα ήθελα να επαναλάβω ότι η πρόταση είτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε της εισηγήτριας δεν απειλεί την αρμοδιότητα που έχει το κάθε κράτος μέλος να φορολογήσει. Αντιθέτως, δίνει περισσότερη ευελιξία στις υφιστάμενες αρμοδιότητες του κράτους μέλους. Σημειώνω ότι είναι σημαντικό ότι δεν ε, επιβάλλουμε εμείς τι πρέπει να γίνει με ζητήματα που αποτελούν μέρος της εθνικής αρμοδιότητας των κρατών μελών. Αντιθέτως, αυτά είναι αυτά που έχουν την ευθύνη να προσδιορίσουν τα συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής που επιθυμούν να υιοθετήσουν στο επίπεδο αυτό. Καλωσορίζω το γεγονός ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποσκοπεί στο να αντιμετωπίσει κάποιες από τις προκλήσεις ε, κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα ε, σε ό,τι έχει να κάνει με τις αδικές μεταφορές με την πρόταση της Ευρωβινιέτας, του Ευρωπαϊκού Τέλους Κυκλοφορίας. Οι περισσότερες αλλαγές, τροποποιήσεις ή ε, τροπολογίες θέλουν να ελαφρύνουν το επιπρόσθετο διοικητικό κόστος είτε για το κράτος είτε για τον φορέα εκμετάλλευσης των οδικών μεταφορών. Αυτό είναι το μήνυμα που έχω να σας εκφράσω εκ μέρους της συναδέλφου κυρίας Τίρντρε Κλούινε. Σας ευχαριστούμε κύριε Βαντεκάμπ για την πολύ καλή ανάγνωση του μηνύματος αυτού. Τα καταφέρατε να το αναγνώσετε. Να δώσουμε το λόγο τώρα στον κύριο Χέρτουγκ που εκπροσωπεί την κυρία Ταμπαντέλ. Και εγώ βρίσκομαι στην ίδια θέση, κυρία Ταμπαντέλ, δεν μπορούσα να βρίσκεται εδώ σήμερα. Θα σας διαβάσω λοιπόν τη θέση της ε, για το κείμενο αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι ω και εισηγήτρια των σοσιαλιστών για το αρχαίο αυτό, συμφωνώ με τι αρχέ τη Κομισιόν ότι η φορολόγηση θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τη χρήση των υποδομών, παρέχοντα ταυτόχρονα κίνητρα για πιο καθαρέ και πιο αποτελεσματικέ ε, ε λειτουργίε. Καλωσορίζω την πρόταση τη Κομισιόν για περαιτέρω βήματα. Συμφωνώ, χρειαζόμαστε περισσότερα εργαλεία για τις επενδύσεις, για τις υποδομές και για τη μείωση της συμφόρηση τη συγχωρήπανσης ε, και της μόλυνσης. Το κείμενο όπως έχει αυτή τη στιγμή δεν καλύπτει αυτές τις ανάγκες, δεν αφορά την πραγματική χρήση υποδομών ενώ θα μπορούσαμε στο μέλλον να χρησιμοποιήσουμε πολύ αποτελεσματικά τα διόδια βάση απόσταση. Έχω δύο προτάσει για μια πιο ισόρροπη προσέγγιση. Πιστεύω ότι η μείωση των ελάχιστων επιπέδων φορολόγηση για τα ε, βαρέα ε, ε, οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων θα μπορεί να λαμβάνει χώρα μόνο εφόσον λαμβάνουμε υπόψη, απόψη την απόσταση στη φορολόγηση. Έτσι αποφεύγονται διπλές φορολογήσεις και τυχόν ανισορροπίες σε τοπικούς προϋπολογισμούς σε ορισμένες χώρες. Και δεύτερον, όσον αφορά το χρόνο, για αυτή τη μείωση θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή για το πώς θα επηρεάσει τις διοικήσεις κάθε κράτου Συνεπώς, η πρόταση της Κομισιόν για μείωση σε μόνο πέντε χρόνια δεν φαίνεται ρεαλιστική, αφού δεν έχουμε σαφή εικόνα του ποια οχήματα θα υποβάλλονται σε τέλη και μπορεί να επηρεάσει δυσανάλογα κάποιες χώρες που βασίζονται στις οδικές μεταφορές. Δεδομένων αυτών, θεωρώ ότι πρέπει να επιτύχουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της εισαγωγής ε, φορολόγησης βάσει απόστασης, μείωσης των οχημάτων και του καλύτερου χρονοδιαγράμματος ε, κυκλοφορίας ε, και πραγματοποίηση της αλλαγής. Ευχαριστούμε κύριε Ερτούγκ. Κύριε Ρίκε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Όπως είπε και ο Βίμ, ελάχιστες ήταν οι τροπολογίες ε, έχουμε παραμείνει πιστοί στο κείμενο της Κομισιόν σε μεγάλο βαθμό. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι φιλοσοφικά ευθυγραμμιζόμαστε με την Ευρωβινιέτα. Κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό, πέραν των όσων υπόθηκαν για τη σχετική ελευθερία των κρατών μελών ε, δεδομένης επικουρικότητας ε, και της ανταγωνιστικότητας. Ε, σημαντικό λοιπόν είναι η δυνατότητα εναρμόνισης, τεχνολογικής εναρμόνισης κυρίως χωρίς ωστόσο ε, να ξεχνάμε το πολύ περίπλοκο πρόβλημα που έχει πολλές προσφορές ε, και που έχει αφαιθεί να εκκρεμεί με αυτή την τροπολογία του κανονισμού. Οι πολλές λοιπόν τροπολογίες δεν αντιστοιχούν σε δικές μας θέσεις αλλά τις υποστηρίζουμε δεδομένου ότι θέλουμε ευρεία ε, υποστήριξη για αυτό το κείμενο, διότι σε γενικέ γραμμέ ευθυγραμμίζεται με την Ευρωβινιέτα που ε, σέβεται νομίζω την αρχή τη επικουρικότητα, αλλά και το άνοιγμα, την απελευθέρωση, ε, χωρί να ξεχνάει την επικουρικότητα των κρατών μελών. Η ισορροπία μα μας φαίνεται ικανοποιητική και δεν και το μέλλον για αυτά τα θέματα, όχι μόνο πολιτικά, αλλά ούτε μόνο κανονιστικά αλλά και σε επίπεδο τεχνολογικό. Το κείμενο αυτό λοιπόν θεωρώ εγώ δεν θα, ε, δημιουργήσει προβλήματα για την ομάδα μας. Ευχαριστούμε κύριε Ρικέ. Κύριε Ντάλον, δείχτε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και πάλι ε, θα πω λίγα λόγια στο όνομα του συναδέρφου Κράμερ για την πρόταση αυτή. Το σημαντικότερο για μας είναι να έχουμε φορολογία οχημάτων που να διασφαλίζει ένα βιώσιμο σύστημα μεταφορών. Με τη φορολόγηση των οχημάτων λοιπόν θα πρέπει αφενός ε, η φορολογία να συνδέεται με το ε, βάρος ώστε η φορολογία να μην ευνοεί τα βαρέα οχήματα αλλά να ευνοεί τα όσο γίνεται ε, πιο ελαφρά οχήματα. διότι με τα βαρέα οχήματα έχουμε περισσότερες εκπομπές και περισσότερη φθορά των οδών. Θέλουμε λοιπόν η φορολογία να προωθεί, τα, να ευνοεί τα ελαφρά οχήματα. Και επίσης ε, να δημιουργήσουμε κίνητρο στους ε, πελάτες να αγοράζουν οχήματα ε, φιλικά όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος και να ενθαρρύνουμε και τις ε, έρευνες ε, και την παραγωγή οχημάτων που να μπορέσουν να συμβάλλουν σε μια πράσινη μεταρρύθμιση στον τομέα των μεταφορών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Κύλωναν, Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. θα ήθελα να μεταφέρω ε, τους χαιρετισμούς ε, της σκιώδους εισηγήτριάς μας ε, που είναι πολύ ικανοποιημένοι με τη συνεργασία και με τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Να δούμε ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστούμε κυρία Κιλόνεν, κύριε Πίτερ Λούγκρεν. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Σημαντικό είναι να είναι φιλικές προς το περιβάλλον οι μεταφορές. Εάν κοιτάξουμε τα πολύ μεγάλα ε, οχήματα, ε, ε, έχουμε τα οχήματα 24, 24 μέτρων στην Σουηδία, τα οποία ε, ναι μεν ε, είναι πιο βαριά αλλά είναι πιο ε, φιλικό προς το περιβάλλον να μπορούμε να φορτώσουμε όσο γίνεται περισσότερα σε ένα φορτηγό και να μειώσουμε τον αριθμό των φορτηγών στον δρόμο. Οπότε τα βαρέα οχήματα τελικά είναι πιο φιλικά στο περιβάλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λούνκρεν. Κύριε Λεζοά, εκ μέρους της Επιτροπής, η άποψή σας για αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπενθυμίζουμε το στόχο της πρόταση. Δεν θέλουμε να υποχρεώσουμε τα κράτη-μέλη να μειώσουν το φόρο. Θέλουμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να τον μειώσουν ω κίνητρο για να καταλήψουν τη φορολόγηση και να περάσουν σε οδικές χρεώσεις, ε, σε διόδια δηλαδή. Σημειώνουμε ότι θέλει απλούστευση ο εισηγητή. Ε, εμείς προτείνουμε μείωση του επίπεδου των φόρων σε πέντε βήματα. Και σκοπός του συγητή είναι να απλουστεύσει τα πράγματα και να έχουμε μόνο ένα βήμα. Θα έλεγα γιατί όχι, αλλά μετά δεν καταλαβαίνουμε γιατί η συγγήτρια σε μια τροπολογία δίνει τη δυνατότητα να μειωθεί ο φόρος μόνο πέντε χρόνια μετά από την θέση σε ισχύ της νέας οδηγίας. Αφού στόχος είναι η απλούστευση, ναι, συμφωνούμε, αλλά θα πρέπει να δώσουμε και μια ευελιξία στα κράτη-μέλη να μειώσουν το επίπεδο των φόρων το συντομότερο δυνατόν. Σε ένα βήμα από τη θέση σε ισχύ της νέας οδηγίας και όχι πέντε χρόνια μετά από τη θέση σε ισχύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Βαντεκάμπ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι οι σκιώδεις εισηγητές έκαναν πολύ αξιοπρόσεκτες παρατηρήσεις. Θα τις διαβιβάσω στην Τίρτρε. Θα διαβιβάσω και τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κατά πώς θα έχουν προσέγγιση σε ένα ή σε δύο βήματα, σε ένα ή σε δύο στάδια. Και θα επανέλθουμε με τα αποτελέσματα των περαιτέρω διεργασιών μας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ψηφοφορία για την έκθεση αυτή θα λάβει χώρα στις 24 Μαΐου στις 9 το πρωί. Συνεχίζουμε με την έκθεση του κυρίου Μασιμιλιάνο Σαλίνη που δεν είναι εδώ και ο κύριος Βιμ Βάντερ θα εκπροσωπήσει τον κύριο Σαλίνη για άλλη μια φορά. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος κύριος Σαλίνη δεν μπόρεσε να έρθει διότι φαίνεται ότι υπάρχουν απεργίες στην Ιταλία που παρακόλλησαν τη μεταφορά του, την έγκαιρη μετάβασή του στην Επιτροπή μας. Και γι' αυτό για άλλη μια φορά θα αναγνώσω το κείμενό του για να δουν οι συναδέλφοι και οι σχεδόντες εισηγητές κατά πόσο συμφωνούν με την προσέγγιση του. Η πρόταση αναδιατύπωσης για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεοδιοδίων και τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για μη καταβολή οδικών τελών στην Ένωση υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Μάιο και έχουμε και την αναθεώρηση της οδηγίας, η οποία αποσκοπεί σε δύο επιδιώξεις. Από τη μία καλύπτεται το ζήτημα της έλλειψης διαλειτουργικότητας των συστημάτων τηλεδιοδίων. Στην αδιατύπωση δουλεύουμε έτσι ώστε η διαλειτουργικότητα των συστημάτων να καταστεί πιο αποτελεσματική, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει τώρα, διότι τώρα έχουμε διαφορετικά συστήματα τηλεδιοδίων τα οποία δεν μπορούν να ε, συνομιλήσουν μεταξύ τους. Επομένως, ε, όλα αυτά πρέπει να διευκολυνούν την διασυνοριακή ε, κινητικότητα και την ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων και αγαθών. Και θα επιτύχουμε το σκοπό αυτό προσδιορίζοντας με σαφήνεια το ρόλο του κάθε παράγοντα, του κάθε φορέα που παρεμβαίνει, του κάθε χρήστη, έτσι ώστε ε, να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για το πώς θα χρησιμοποιείται το σύστημα αυτό. Από εκεί και πέρα, η οδηγία λύνει το πρόβλημα των ε, ελληματικών πληρωμών. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει ανταλλαγή ε, δεν μπορεί να υπάρξει ανταλλαγή των στοιχείων της πινακίδας κυκλοφορίας και τα λοιπά των οχημάτων ε, με σκοπό να εισπραχθούν τα διόδια μεταξύ των κρατών μελών. Δεν μπορεί να υπάρξει ανταλλαγή και αυτό είναι απώλεια 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Επομένως, ε, καλωσορίζουμε το γεγονός ότι δημιουργείται αυτή η νομική βάση, την προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αναδιατύπωση και θα λυθεί το πρόβλημα αυτό. Για να πετύχουμε τους φιλόδοξους αυτούς στόχους, Συζητήσαμε με τους κοιόδης εισηγητές και καταλήξαμε σε οκτώ συμβιβαστικές τροπολογίες για τα πιο σημαντικά ζητήματα της οδηγίας και ήδη έχει βρεθεί συμφωνία για τις περισσότερες από αυτές ειδικότερα για τη συμβιβαστική τροπολογία που έχει να κάνει με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη συχνότητα της υποβολής των στοιχείων αναφοράς. Συνεχίζεται η συζήτηση για το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας και εκεί συμπεριλαμβάνεται το ΟΥΒΑ για την αστική κινητικότητα και το ρόλο των συστημάτων ANBR. Σε κάθε περίπτωση είμαι βέβαιος ότι θα βρούμε συμφωνία και ε, θα πετύχουμε συμφωνία και πάνω σε αυτά τα ζητήματα στην τελευταία συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών την επόμενη Τετάρτη. Έρχομαι τώρα με ένα νέο σχέδιο πρότασης που έχει συμπεριλάβει τις περισσότερες προτάσεις των σκιωδών εισηγητών και μάλιστα το συντομότερο δυνατό και γι' αυτό δεν έχουμε και σαφή κείμενο ακόμα. Σε αυτές τις συμβαστικές τροπολογίες έχουμε μια καινούρια για τα εδάφια που έχουν να κάνουν με την απόφαση. Θα προσθεθεί αυτό. Για άλλη μια φορά θέλω να σας ευχαριστήσω για την επικοδομητική συνεργασία που επέδειξαν όλοι οι συνάδελφοι καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής. Ε, συναδελφοί, ε, ο φαινόμενος κ. Βαντεκάμπα ε, προσθέτει τον πληθυντικό. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Βίμ Βάντερ Η κυρία Σενάλοβα έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη στάση του, για την επικοδομητική του δουλειά. Πράγματι σας επιβεβαιώνω ότι εμείς καταφέραμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία σε ό,τι έχει να κάνει με τις περισσότερες τροπολογίες. Θέλουμε να δημιουργήσουμε τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες για την θέσπιση ενός ηλεκτρονικού συστήματος το οποίο να έχει ε, διαλειτουργικότητα. Πολλές ε, τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και δεν θα είναι στο παράρτημα αυτές, αλλά θα είναι στο διατακτικό του κειμένου. Και θέλουμε να συμπεριληφθεί και το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης των πινακιδών κυκλοφορίας. Γιατί και αυτό θα βελτιώσει τα μάλα το σύστημα τηλεδιοδίων στις ζώνες χαμηλής εκπομπής αερίων ε, του φαινομένου θερμοκηπίου. Σε κάθε περίπτωση θα έχουμε και άλλη συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών και θα μιλήσουμε και για την ανταλλαγή, τη διασυνοριακή ανταλλαγή των προσωπικών δεδομένων. Βεβαίως και περιμένουμε τις βασικές σκέψεις, τις τελευταίες ιδέες και τροπολογίες που έχουν οι σκιώδεις να υποβάλλουν. Ε, πέρα από αυτά όμως έχω την αίσθηση και το ελπίζω ότι η συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας θα μας βοηθήσει ιδιαίτερως να ε, καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριος Φανίλτεμπεργκ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Κυρία Πρόεδρε, λυπάμαι που έχασα ε, τη συζήτηση, αλλά φαίνεται να τρέχετε τόσο πολύ με την ημερήσια διατάξη σήμερα που έχασα κάποια κομμάτια τη συζήτηση. Ζητώ συγγνώμη. Σε κάθε περίπτωση, όλοι γνωρίζουμε, πιστεύω, τη συζήτηση αυτή μεταξύ ε, εισηγητή και σκιωδών. Δεν υπάρχουν μυστικά. Εργαζόμαστε σε πολύ θετικό περιβάλλον. Έχουμε κάνει και τις προτάσεις που πιστεύω ότι θα είναι καλές όσον αφορά την οδηγία θα παρέχουν μεγαλύτερη ε, νομική ασφάλεια. Είναι σημαντικό. Έχουμε κάνει προτάσεις και για τους παροχούς υπηρεσιών που πιστεύω θα βοηθήσουν. Ένα κομμάτι του Κοινοβουλίου δεν ε, ακούει αυτά που εγώ θεωρώ πολύ σημαντικά. Το ότι πρέπει να οι τεχνικές απαιτήσει να μπορούν να τροποποιηθούν με ε, της πράξη εκτελεστικές πράξεις παρά να περιλαμβάνονται στο κυρίως κείμενο της οδηγίας διότι αυτό θα χρειαζόταν πολύ καιρό για οποιαδήποτε επικαιροποίηση σε περίπτωση που υπάρχουν νέε τεχνολογίε στην αγορά. Πρέπει να μπορεί κανεί να επικαιροποιήσει γρήγορα την νομοθεσία του. Γι' αυτό εγώ ήθελα κατ' η εκτελεστική πράξη. Κάποιοι σκιώδει εξέφρασαν δισταγμού, αλλά είναι πολύ σημαντικό θέμα αυτό κατά την άποψή μου. Γενικότερα είμαι πολύ ικανοποιημένο που πολλοί σκιώδει και ο εισηγητή έχουν δει θετικά πολλέ από τι συμβαστικέ και διασφάλισαν η αυτόματη αναγνώριση πινακίδων κυκλοφορία να συμπεριληφθεί. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, ειδικότερα ε, για τα διόδια. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η βάση ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα λαμβάνει πράγματι τα χρήματα. Επίσης είναι σημαντικό και σε διασυνοριακή βάση να μπορεί κανεί να γνωρίζει ότι μπορεί να συγκεντρώσει να συλλέξει τα έσοδα από του ξένου οδηγού. Είναι πολύ τεχνική φύση αυτό το αρχείο, θα το έχουν καταλάβει οι συνάδελφοι. Οι συζητήσεις θα γίνουν αυτή την εβδομάδα, αλλά ελπίζουμε ότι η τελευταία μα συνάντηση με τους Κιώδη θα είναι αυτή την εβδομάδα και ότι θα μπορέσουμε να ψηφίσουμε 24 Μαου όπω έχει προβλεφθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Νταλούντε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή για την δουλειά του καθώς ε, και ευχαριστώ για την καλή συνεργασία μεταξύ των σχεδόν εισηγητών. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Μπορεί να φαίνεται τεχνικό διότι πολλές ε, χώρες ε, και πόλεις εισάγουν διαφόρων ειδών τέλη στου δρόμους και δεν υπάρχει διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων αυτών για να διευκολύνεται ο οδηγό. Αλλά στην ε, σημερινή κοινωνία μπορεί να ζούμε σε μία πόλη, να δουλεύουμε σε άλλη. Γι' αυτό είναι σημαντική η διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων. Η πρόταση αυτή επικεντρώνεται στο ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιούνται μόνο για τους συγκεκριμένους στόχους και θα πρέπει να είναι δυνατή η πολυτροπικότητα ώστε στο μέλλον να ενθαρρύνουμε τους πολίτες να χρησιμοποιούν λιγότερο το αυτοκίνητό τους και να προτιμούν άλλους τρόπους μεταφοράς. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νταλούντε. Κυρία Κιλόνεν, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συνάδελφοι, Ο σκιώδης εισηγητής ε, της ομάδας μας ε, στέλνει τους ε, χαιρετισμούς τους προς την ομάδα. Ήταν εξαιρετική η συνεργασία και θα ήθελε απλά να αναφέρει ότι οι συμβιβαστικές προτάσεις φαίνεται να μπορούν να γίνουν αποδεκτές από εμά και νομίζω ότι αυτό αποτελεί πολύ καλή απάντηση προς τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητέ. Μπορεί να μην είναι τέλεια η λύση, αλλά βρίσκεται πολύ κοντά νομίζω στην τελειότητα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Κίλωνεν. Ο κύριος Λούντκρεν. Ναι, όλοι σκέφτονται το περιβάλλον, πολύ ωραία ακούγεται αυτό. Νομίζω ότι είμαι το μόνο μέλος όμως της Επιτροπής μας που κινείται που μετακινείται με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Άλλα λέμε, άλλα κάνουμε. Πώς ε, λοιπόν θα ποντάρουν οι απλοί άνθρωποι σε, στην τεχνολογία αυτή, ναι, αν δεν τη χρησιμοποιούμε εμείς εδώ στην Επιτροπή μας. Ε, και όταν μιλάμε για αναγνώριση των πινακίδων κυκλοφορίας, θα ήθελα να αναφέρω ότι τα, οι πλαστές πινακίδες αποτελούν σημαντικό πρόβλημα ε, στον τομέα των μεταφορών. Ε, μάλιστα, ε, μπορεί να αγοράσει κανείς πλαστές πινακίδες. Πολλούνται σουηδικά φορτηγά και δύο ώρες αργότερα έχουν ξένες πινακίδες. Όσο ωραία λοιπόν και αν μιλάμε για το περιβάλλον και το ότι θα πρέπει όλοι να πληρώσουμε, τη στιγμή που ε, κυκλοφορούν ένα σωρό αυτοκίνητα με πλαστές πινακίδες για τα οποία δεν έχουμε ε, έλεγχο επειδή δεν υπάρχει η διεθνής βάση δεδομένων που να μπορεί να ελέγξει η αστυνομία, ε, τότε δεν έχει νόημα όλο αυτό που λέμε. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μία συσκευή αναγνώρισης ώστε και η αστυνομία να μπορεί να αναγνωρίζει τις πλαστές πινακίδες διότι αλλιώς τελικά πάλι οι απλοί πολίτες θα πληρώνουν το λογαριασμό που θα πρέπει να πληρώνουν άλλοι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Λόντκρεν. Η Κομισιόν. Κύριε Λεζό, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Από την τελευταία ανταλλαγή πληροφοριών που είχαμε τον Μάρτιο, νομίζω οι εξελίξεις ήταν πολύ καλές, όχι μόνο στο Κοινοβούλιο, αλλά και στο Συμβούλιο. Την περασμένη εβδομάδα συνεδρίασε για τελευταία φορά η ομάδα εργασίας. Έχει προχωρήσει το κείμενο πολύ και είναι πολύ πιθανό να εγκριθεί από το Συμβουλίο Υπουργών στις 7 Ιουνίου. Επί της ουσίας, δύο παρατηρήσεις. Δουλέψαμε πολύ με τον εισηγητή και με τη γραμματεία της Επιτροπής Μεταφορών για να πετύχουμε το σωστό σημείο ισορροπίας μεταξύ των διατάξεων που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην οδηγία και τα μη απαραίτητα στοιχεία που μπορούν να εφαρμοστούν και να συμπεριληφθούν στην εφαρμοστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένα παράδειγμα συμπερίληψη στην οδηγία είναι αυτό που έχει να κάνει με το πάροχο. Πρέπει να αναγνωριστούν όλα αυτά τα στοιχεία και να συμπεριληφθούν στην έκθεση που θα ψηφιστεί για να αποτελέσει αυτή η έκθεση τη βάση για τον τριμερή διάλογο με το Συμβούλιο. Τώρα, μια δεύτερη παρατήρηση δική μου, πιο επικριτική, έχει να κάνει με την τροπολογία του εισηγητή για να αποκλειστεί ε, η αυτόματη αναγνώριση των πινακιδών κυκλοφορίας, το ANPR. Εμείς είμαστε κατά ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί θεωρούμε ότι το σύστημα συμβάλλει ιδιαίτερος στην καταπολέμηση των απουσιών πληρωμών είναι χαμένη ευκαιρία εάν δεν το περιλάβουμε στη διαλειτουργικότητα. Είναι πραγματικά κρίμα. Ε, καλούμε τον εισηγητή να επανεντάξει αυτή τη τεχνολογία στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Α, κατά τα λοιπά και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είμαστε στο σωστό δρόμο και το επόμενο βήμα είναι η υπερψήφιση στην Επιτροπή Μεταφορών. Ευχαριστώ κύριε Λεζουά, κύριε Πιμ Βαντερκάμπ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. θα μεταφέρω όλες τις παρατηρήσεις των συνάδελφων των κ. Σαλήνη, ακόμη και αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φυσικά ώστε να τα συμπεριλάβει ε, να συμπεριλάβει και την τεχνολογία. Θα ήθελα, ο κ. Σελήνη να ευχαριστήσει όλους ε, θα πρέπει όλοι να ακούσουμε σωστά όλα τα σχόλια που έχουν γίνει ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι λεπτομέρειες μας γιατί είναι ύψης της σημασίας. Ευχαριστώ πολύ. Υπενθυμίζω ότι η ψηφοφορία για την εκθέση αυτή θα λάβει χώρα στις 24 Μαΐου από τις 9 η ώρα. Λοιπόν, τα κάναμε όλα πολύ γρήγορα. Κανονικά η συνεδρίαση των συντονιστών ε, πρέπει να ξεκινήσει τώρα, αλλά δυστυχώς κάποιοι συντονιστές δεν είναι εδώ. Διακόπτουμε λοιπόν και θα επιστρέψουμε στις 5.30. Ε, ναι. Παραμένει η ώρα. Ευχαριστώ. Τα λέμε μετά. Ή αλλιώ μπορούμε να την κάνουμε νωρίτερα, αν θέλετε. Τι να πούμε, πέντε. Πέντε η ώρα. ο κύριος Τέχνης δεν είναι εδώ. Δεν θα, δεν γίνεται, όχι. Ωραία, θα περιμένουμε λοιπόν μέχρι τις πέντε και μισή. Τα λέμε εκείνη την ώρα.